κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτω ώστε να μην πρέπει να επαναλάβουμε τα υποθέντα σήμερα. Ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση περατώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω κάποια ανακοίνωση. Προάσπιση ασυλίας ενός βουλευτού, του κυρίου Βαλτεμάρ Βαντεβά Τομασεύσκη και αυτό το αίτημα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να προστατευτεί η ανεξαρτησία του κατά τη διάρκεια τη θητεία του ω Ευρωβουλευτή μετά από μια απόφαση που ελήφθη από την βασική Επιτροπή τη Λιθουανία για τη Δεντολογία και απόφαση που τον αφορά. Το διάβημα του κ. Βαντεμάρ Τομαζεύσκη υποστηρίχθηκε από πολλού Ευρωβουλευτέ και εν εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφο 3 του εσωτερικού κανονισμού αυτό το αίτημα απεστάλλει στη νομική επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση Σκότα για την ε, ε στρατηγική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να ακολουθηθεί και σχετική έκθεση. Θα ξεκινήσω λοιπόν δίνοντα στον κύριο Σκοτά, τον Τζαν Κάρλο Σκοτά, το λόγο για ένα τετράλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τη σοβαρή κρίση που ζει η Ευρώπη, και στον γεωργικό τομέα, μία από τι απαντήσει που μπορεί να δώσει η αγροτική αγορά είναι να βασιστεί στην ποιότητα των προϊόντων. Πιστεύω ότι μια καλή ποιοτική πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να δώσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία των περιφερειών τη Ευρώπη, που πολύ συχνά είναι η μόνη δυνατότητα για ανάπτυξη αυτέ τι περιοχέ. Για πολλέ περιοχέ τη Υπέθρου που είναι με νυχτική θέση, με περιορισμένε εναλλακτικέ δυνατότητε παραγωγή. Υποστηρίζοντα λοιπόν τη γεωργία σε αυτέ τι μειονεκτούσε περιοχέ, δημιουργούμε οικονομία και θέσει απασχόληση στι περιοχέ αυτέ. Πέραν αυτού, μια μελλοντική πολιτική ποιότητα θα πρέπει να βασίζεται βασίζεται και στι δυνατότητε που έχει μια σύγχρονη γεωργία που είναι δυναμική και πλούσια και με ποικιλομορφία όπω αυτή είναι η ευρωπαϊκή γεωργία που μπορεί να προσφέρει όχι μόνο τρόφιμα ύψης της ποιότητας αλλά και υπηρεσίε που κοινοφελείς για μια κοινωνία που συνεχώ εξελίσσεται. Στην έκθεσή μου υπογράμμισα τη σημασία που έχει να κρατήσουμε ξεχωριστά τα τρία συστήματα καταχώρηση των ενδείξεων γεωγραφική προέλευση και έχω και το παράρτημα που δείχνει τι γίνεται στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, περιοχές Εκπροσωπούνται εκεί παραδόσει, ιστορία, το γούστο και οι γνώσει οι αποκλειστικέ ε, που έχουν περάσει, έχουν διαδοθεί με την πάροδο του χρόνου. Θα, εάν έχουμε τον DOP και HGP, τα δύο συστήματα ξεχωριστά, ε, θα πρέπει να λάβουμε έτσι τι διαφορέ που υπάρχουν όσον αφορά τη μορφή και την ένταση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ του προϊόντο και τη περιοχή παραγωγή. Οι καταναλωτέ πολύ συχνά συγχαίουν την ένδειξη ε, τον τόπο με τον οποίο είναι η κατεργασία του προϊόντο με την προέλευση του αρχικού προϊόντο και πολύ συχνά δεν γνωρίζουν το πώ λειτουργεί η όλη τροφική αλυσίδα. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι μόνο η ένδειξη υποχρεωτική του τόπου παραγωγή των πρώτων υλών, των πρώτων προϊόντων μπορεί να δώσει στον καταναλωτή την πραγματική γνώση όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος το οποίο αγοράζει. Λοιπόν, ε, υπόκειται σε έναν κύκλο παραγωγής που μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του το προϊόν σε σχέση με την ποιότητα και την πιστιστική ε, ασφάλεια, την ασφάλεια του τροφίμου. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε αυτό που παράγεται και αυτό που καταναλώνουν οι πολίτε μα που μα ψήφισαν. Άλλα δύο θέματα που θεώρησα ότι είναι σημαντικά και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή μου είναι η σημασία που έχει να υπάρχει εντατικοποίηση τη εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες ετικέτες που φθήθενται και στις εγγυήσει που δίνουν αυτές οι ετικέτες και τα σήματα. Και στα εθνικά μητρώα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η διεθνή αναγνώριση του συστήματο του ΠΟΕ των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι θεμελιώδου σημασία αν θέλουμε να προστατεύσουμε από παραποίηση τα διάφορα ποιοτικά μας προϊόντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τσόλοφ για την, ε, για την παρουσία του, υπενθυμίζοντα τη σημασία που έχει μια επαρκή προστασία των διαφόρων συστήματων ποιοτική εξασφάλιση που έχουμε στην οικονομία. Η οικονομία τη υπαίθρου που, των περιοχών που μειονεκτούν μπορεί να βοηθηθεί αν βοηθήσουμε το γενικό τομέα που διαφυλάσσει όλα αυτά τα ε, τυπικά προϊόντα των διαφόρων αυτών περιοχών και έτσι οι πληθυσμοί που παράγουν τα προϊόντα παραμένουν επιτόπου που διαφορετικά θα είχαν εγκαταλείψει την περιοχή τους θα πρέπει βέβαια να σεβόμαστε το περιβάλλον, την ύπεθρο και όπου είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε και μια τουριστική οικονομία και είναι γαστρονομική οικονομία που συνδέεται με τι διάφορε περιφερειακέ διαφορέ που υπάρχουν και αντικατοπτρίζουν την ιστορία και την ποικιλομορφία τη Ευρωπαϊκή Ενέση. Ευχαριστώ του συναδέλφου την υποστήριξη που μου έδωσαν στην Επιτροπή Γεωργία και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει το ίδιο αύριο κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ κύριε Σκότα. Να δώσω το λόγο τώρα ονόματα της Επιτροπής στον κύριο Τσιόλος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σκοτά, κυρίε και κύριοι, θεωρώ ότι το κεντρικό στοιχείο που δίνει προσωπικότητα στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο σε διεθνές επίπεδο είναι ακριβώς η πολιτική ποιότητας και ποικιλότητας και γι' αυτό η πολιτική ποιότητα στον γεωργικό τομέα θα είναι μία από τις κατά διάρκεια της ε, θητείας μου. Η ποιότητα μετά την αναθεώρηση της ε, ΚΑΠ ε, μετά το 2013. Η ποιότητα. βλέπουμε ότι οι παραγωγοί αντιδρούν στις απαιτήσει των καταναλωτών και επίσης θα μπορούσε η ποιότητα αυτή να προωθήσει στη διεθνή αγορά τα προϊόντα της ε, αγροτικής ε, βιομηχανίας. Θα πρέπει να ενταχθούμε σε ένα σαφές ε, πλαίσιο δομημένο, κατανοητό από τους κατανοητές και επαρκές. Ο στόχος μου στην πολιτική ποιότητα είναι να είναι πιο προσιτή και για τους παραγωγούς που θα πρέπει να ωφεληθούν αλλά και για τους καταναλωτές χωρίς να χάσουμε την ουσία και το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής. Η πολιτική ποιότητα σημαίνει μια εξασφάλιση για το καταναλωτή. Ταυτόχρονα όμως και μια προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς. Συμφωνώ με τον κύριο Σκότα από αυτό. Συμβάλλει στην διατήρηση της ε, διαφοροποίησης των παραγωγών και της αγωνιστικότητά τους γιατί μία ε, γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να πουλάει τα προϊόντα της είναι ανταγωνιστική. Εάν δει από αυτό είναι ανταγωνιστική. Και εάν πολλά προϊόντα με υψηλή προστάμενη αξία είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική. Ακόμα και αν καμιά φορά πρόκειται για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική ποιότητα σε ορισμένου τομεί θα μπορούσε να και περιφέρειε θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αύξηση τη αγνωστικότητα των περιφερειών αυτών. Θεωρώ ότι η πολιτική ποιότητα, η ανάπτυξη των τοπικών αγορών και η καλύτερη επαφή καταναλωτών και παραγωγών θα μπορούσε να δώσει κίνητρα για την αύξηση της αναγνωστικότητας ωραίων προϊόντων που δεν είναι και τόσο έντονη η παρουσία του στην αγορά οι παραγωγοί προσπαθούν να προσφέρουν ασφαλή προϊόντα με τεχνολογίες που σέβονται την ευημερία των ζώων και το περιβάλλον. Θεωρώ ότι είναι καλό να βοηθήσουμε με την σήμανση των προϊόντων αυτών και το αναφέρει και η έκθεση. Αυτός ο σχετισμός μεταξύ των προτύπων που τηρούν οι ε, παραγωγή για την πολιτική ποιότητα και την σήμανση θα είναι ένα θέμα και τη συζήτηση που θα κάνουμε για το μέλλον της ε, αγροτικής πολιτικής μετά το 2013. Θα πρέπει να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε τα μέσα μας για την πολιτική και όσον αφορά τους καταναλωτές, αλλά κυρίως τους καταναλωτές σε διεθνές επίπεδο. Το σύστημα ποιότητάς μα θα μπορούσε να προωθήσει το σύστημα της αγροτικής μας πολιτικής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κατάλληλη στιγμή στην οποία παρουσιάζεται η έκθεση Σκότα. Ε, ξέρετε ότι η Κομισιόν προετοιμάζει μία έκθεση μέχρι τα τέλη 2010 για την ποιότητα των γεωρικών προϊόντων. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει διάφορα θέματα, ιδέες, προτάσεις και οπωσδήποτε θα αντιλέγω υπόψη κατά το δυνατόν όταν θα έρθω ενώπιον ημών με τις νομοθετικές προτάσεις θα την έχω μελετήσει. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τα μέλη της Αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου που εργάστηκαν για την έκθεση αυτή και με χαρά θα ακούσω τις απόψεις και τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παράδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο η κυρία Ραντ Καρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σήμερα Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκοτά για την εξαίρετη διάθεση που επέδειξε για συνεργασία για την έκθεση αυτή. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα και για τους υπόλοιπους από τις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες να συνεργαστούμε μαζί του. Και είμαστε περήφανοι για την πρόταση που θα προτείνουμε σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και είμαστε περήφανοι γιατί πιστεύω ότι στηρίζουμε με την έκθεση αυτή την ποιότητα και τις ορεινές περιοχές και τις περιοχές της Υπέθρου. Είναι μια παράδοση για την Ευρώπη οι περιοχές αυτές, αλλά επίσης ε, μας προσφέρουν πλούτο και θέσεις απασχόλησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης και ανεργίας σε πολλές χώρες μέλη. Επίσης, ε, μας ικανοποιεί το γεγονός ε, ότι η θέση αυτή της Επιτροπής Γεωργίας είναι υπέρ της ποιότητας στον ανώτατο βαθμό. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στις ονομασίες προέλευσης και στις ε, ενδείξεις προέλευσης. Δεν πρέπει να υπάρξει μείωση της ποιότητας. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε την κοινωτική παραγωγή. Χαίρομαι για τόσα μας είπε ο Επέτροπος. Είναι χαρά για μας να τον ακούμε να στοιχηματίζει υπέρ του μέλλοντος στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ελπίζουμε να ακούσει και τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα φανεί αύριο με την ψηφοφορία. Τέλο, ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο και να αποφασίζει πράγματα όπω είναι για παράδειγμα ε, τα πρότυπα εμπορία. Θέλουμε οι διορθώσει που γίνονται στην αγορά να αλλάξουν. Θέλουμε και εμείς να στοιχηματίσουμε υπέρ της ασφάλειας της διατροφικής, της ποιότητας, και της ε, σωστής παραγωγής. Οι κοινοτικές προδιαγραφές και η ποιότητα της ε, παραγωγής τροφίμων από την κοινότητα είναι πολύ βασικό και πρέπει αυτό να το δούμε και μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους παραγωγούς μας με διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των ομάδων τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τζοβάνι Λαβία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εν ονόματι της ομάδας του ΕΛΚ τον κύριο Σκοτά, τον εισηγητή για τη λαμπρή δουλειά που έκανε και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ποιοτικέ πολιτικές οι πολιτικές ποιότητες μάλλον εκτός του να δώσουν μια προστιθέμενη αξία σε αυτά που προσφέρουν στους καταναλωτές έχουν και μεγάλη σημασία για εκείνο που μπορούν να δώσουν στους ε, παραγωγούς. Όπως σημειώνεται όλοι, ο ανταγωνισμός μπορεί να ε, εφαρμοστεί ποικιλόμορφα σε διάφορες αγορές. Σε μια μεγάλη χώρα, όπου είναι η Ευρώπη, σε μια τόσο σύνθετη, πολυσύνθετη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται όμως από υψηλό κόστος παραγωγής έναντι του ανταγωνισμού, θα είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις τιμές και ο ανταγωνισμό θα μπορεί να διεξαχθεί μόνο μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων. Και από αυτή την οπτική γωνία της διαφοροποίησης θα πρέπει να δούμε την πολιτική ποιότητα, να μπορούμε να προσφέρουμε και να θέτουμε στην αγορά ένα προϊόν διαφορετικό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το μπορεί με συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να προσφέρεται και ε, παρόλα αυτά και σε χαμηλότερη τιμή εναντί του ανταγωνισμού. Που δεν μπορεί να προσφέρει σε, να προσφέρει σε χαμηλότερη τιμή. Ε, ξεκίνησαν τα κοινοτικά σήματα σαν πείραμα και είδηξαν ότι υπάρχει ανάγκη να κρατήσουμε τη διαφορά μεταξύ γεωγραφικής ενδείξεως ε, και ονομασίας προέλευσης. Και θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε και σε διεθνές επίπεδο και στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο τη θέση μας και να υπερασπιστούμε την πολιτική αυτή των ονομασιών προέλευσης. Ούτως ώστε να αποφύγουμε μία αναπόφευκτη πολιτική ε, ανταλλαγής ισοδυναμίας αν θέλετε των διαφόρων σημάτων που θα ήταν επιβλαβής για τα προϊόντα μας. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την Ζητήσαμε και θα ζητήσουμε και αύριο με ειδική τροπολογία στην ψηφοφορία του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα να αναφέρεται στην ετικέτα η προέλευση της πρώτης ύλη. Όχι μόνο για τα νοπά μη μεταποιημένα προϊόντα, αλλά και για τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν ένα μόνο στατικό. Δηλαδή εκείνα που ουσιαστικά έχουν στην πρώτη τους ύλη το χαρακτηριστικό στοιχείο που εμπεριέχει το τρόφιμο. Ευχαριστώ. Κύριε Λαβή, ο κύριος Ταμπάζντι έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε σε όλες αγαπητοί συνάδελφοι. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πιστεύουν ότι η έκθεση του κυρίου Σκότα είναι πάρα πολύ σημαντική και την κρίνουν πολύ θετικά. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή ε, έχει πολλά καλά σημεία. Παραδείγματος αν το κοινοτικό σήμα. Πολύ δεν καταλαβαίνω αυτό δεν σημαίνει ε, τίποτα άλλο παρά μια εγγύηση ότι τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για την ασφάλεια τροφίμων. Και γι' αυτό μπορούν έτσι να ε, διακριθούν από άλλα προϊόντα, και κυρίως εισαγωγές. Επίσης, έχω να πω ότι χαίρομαι ότι με το πρόσωπο του κυρίου Τσόλο έχουμε έναν επίτροπο σε αυτό το τομέα που υποστηρίζει τις τοπικές αγορές και τους δίνει μια ιδιαίτερη προτεραιότητα. Γιατί ακριβώς ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η ιδιαιτερότητα των προϊόντων αυτών ε, προέλευσης όπως το λέμε. Είναι σωστό λοιπόν να τα σημαίνουμε ξεχωριστά. Χαίρομαι που ο Επίτροπος δεν υποστηρίζει την παλιά άποψη ότι αυτές οι ονομασίες ε, προέλευσης και οι προστατευμένες γεωγραφικές ε, ε, προελεύσει θα πρέπει να συνενωθούν. Φαντάζομαι ότι παρόλο που έχουν λυθεί ακόμα κάποια προβλήματα παραμένουν άλλα άλυτα που ελπίζω ότι θα επιληθούν. Τελευταία παρατήρηση που διάφοροι είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε για τα φρούτα και για τα λαχανικά τις ίδιες αυστηρές διατάξεις όπως οι διαφορετικά προϊόντα αλλά θα πρέπει να μην υπερβάλλουμε σε διακανονισμούς να διακανονίζουν το χάρη τις μπανάνες για το πόσο καμπύλες πρέπει να είναι. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σκότα για την έκθεσή του. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα που συστήνουμε. Δυστυχώς εγώ και οι συνάδελφοι από την Άλντε δεν μπορούμε να στηρίξουμε απόλυτα την έκθεση αυτή χωρίς δύο αλλαγές. Γιατί δεν μπορούμε να στηρίξουμε την παράγραφο 19 γιατί πιστεύουμε ότι είναι ανοησίες για τους γραφειοκράτες της Βρυξέλλες να πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράζουν ίσχες μπανάνες ή αγκουράκια. Για μένα αυτά είναι λάθος. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει την κοινή του λογική και θα στηρίξει τις τροπολογίες εκείνες που είναι κατά τέτοιων ρυθμίσεων και να αφήσουν τον καταναλωτή να αποφασίζει αν θέλει να ψωνίζει και να τρώει ίσχες μπανάνες στις τραβές. Είναι μια απόφαση που πρέπει να την παίρνουν οι καταναλωτές. Ε, η κυρία Φίσερ Μπόλς είχε μιλήσει για αυτές τις προδιαγραφές. Να ξέρετε ότι εμείς συμφωνούμε την προηγούμενη απόφαση. Επίσης θέλουμε κάποιες αλλαγές και στην παράγραφο 16. Εγώ αντιλαμβάνομαι την επιθυμία να υπάρχει ένα γιουρολόγο. Για μένα το σημαντικό είναι να υπάρχει προστιθέμενη αξία και για τους γεωργούς. Να βοηθήσουμε και τους γεωργούς, γιατί αλλιώ δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να πετύχουμε ένα τέτοιο στόχο. Δεν βλέπω γιατί να θέλουν οι καταναλωτές να βρουν αυτό το γυρολόγο. Τέλος για την παράγραφο 62. Αναφέρονται κάποιες ε, κριτικές για το σύστημα ιδιωτικής πιστοποίησης. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό οι αγρότες να μπορούν μέσω τέτοιων προγραμμάτων ποιότητας να δίνουν προστεθέμενη αξία στην παραγωγή τους και πρέπει να το επιτρέψουμε. Θέλω λοιπόν να δω τις αλλαγές αυτές στην αυριανή ψηφοφορία και αν ε, ψηφιστούν αυτές οι αλλαγές τότε εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Λάιον. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Άλεν Σμιθ. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια του Σκοτσέζου συναδέλφου μου, του George Λάιν, παρόλο που δεν συνάδελφο στην ομάδα. Πολλά περιέχει έκθεση, είναι αξιοθαύμαστα και έκανα δύο πράγματα που θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Και υποβάλαμε διάφορε προτάσει, εστιαστώ σε δύο από αυτά μόνο τα σημεία οι, οι καταναλωτές μας θέλουν να ξέρουν πού προέρχεται το τρόφιμο. Αυτό πιστεύουμε. Και η παροχή των πληροφοριών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Αυτό πιστεύουμε. Οπότε η τροπολογία 2 που έχουμε υποβάλει, ακριβώς αυτό. Τροπολογία 4 μάλλον, για τον ομιλητή, αντικατοπτρίζει κάποια δύναμη διατύπωση με ισχυρότερη διατύπωση όπου μπορούν να βάλουμε πληροφορίες για το πού παρήχθη το προϊόν, να το κάνουμε και υποχρεωτικά, γιατί αυτό θέλουν να βλέπουν οι καταναλωτές. Έχουμε και την τροπολογία 3 που ανέφερε συνάδελφο που γράφει να βάλουμε, να επαναφέρουμε πολύ δίσκαμπτους κανόνες, επαχθείς κανόνες όσον αφορά την άμεση πώληση ε, λαχανικών και φρούτων στους ε, καταναλωτές. Είχαμε αποφασίσει πέρσι να ανακληθούν αυτοί οι κανόνες και δεν είδαν μεγάλη διαφορά οι καταναλωτές, αλλά η παραγωγή είδαν τη διαφορά. Η αδίποτε προσπάθεια επαναφοράς των κανόνων θα εμποδίσει και τους μεταποιητές, ε, μάλλον θα δώσει όπλα στα χέρια και των μεταποιητών και των υπεραγορών να καταπιέσουν τους παραγωγούς. Συμφωνώ με αυτά που ο κύριος Λέων για το σήμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ε, Είναι περισσότερο φιλοδοξίε που αφορούν το κοινοβούλιο και όχι αυτό που θέλουν οι καταναλωτές. Και αν δεν είναι λογικό του καταναλωτές, ας μην το κάνουμε και θα πρέπει να αντακατασταθεί με ένα πρόγραμμα για την υποχρεωτική δικαιοθεσία προελεύσεως του προϊόντο Είναι κάτι που θέλουν οι καταναλωτές. Και ελπίζω να υποστηρίξουν αυτέ τι επικοδοκιμητικέ μα τροπολογίε αύριο. Ο κύριο Νίκολσον έχει το λόγο δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ έκθεση. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλε ιδέε, πολλές καλές ιδέες στην έκθεση και συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή τον κύριο Σκότα που λέει πόσο σημαντικό είναι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να προσθέσουν αξία και να μεγιστοποιούν το δυναμικό των προϊόντων τους. Θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να πετυχαίνουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο όσον αφορά τα τρόφιμα της Ευρώπης, ε, το μέγιστο δυναμικό. Θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχυθεί η οικονομία της υπαίθρου. Σχετικά με αυτό χαίρομαι που βλέπω ότι ο κύριος Σκότα αντιμετώπισε το θέμα των, του μέλλοντος των, των σημάτων προέλευσης, ονομασίας προέλευσης ε, και αυτό ωφελεί και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές αλλά η διαχείριση των συστημάτων και εφαρμογή του πρέπει να πλουστευτεί. Αν είμαστε σοβαροί για την αξία αυτών των δύο συστημάτων στο εξωτερικό, θα πρέπει να ασφαλίσουμε ε, και περισσότερη προστασία από τα προϊόντα τρίτων χωρών. Να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα ήθελα να δω περισσότερα προϊόντα από τη δική μου περιοχή να ζητήσουν σήμα πρόελευση, ονομασία προέλευσης ε, και ένδειξη προέλευση ε, Και θα πρέπει να προσθεθεί διαδικασία χορηγήσεως, εγκρίσεως αυτών των σημάτων. Και νομίζω ότι τότε και από την περιοχή μου τη Βόρεια Ιρλανδία θα υποβληθούν περισσότερες αιτήσει αν απλουστευτεί το σύστημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της εκθέσεως που δεν τα υποστηρίζω όμω. Είμαι κατά της εισαγωγή ενό σήματο ευρωπαϊκού για την ποιότητα. Αυτό υποστηρίζω είναι ετικετοθεσία για τη χώρα προελεύσεω. Και νομίζω ότι ένα ευρωπαϊκό σήμα δεν θα είχε νόημα, θα ήταν σπατάλη χρόνου και θα σπαταλούσε και χρήματα και το ίδιο αισθάνομαι και για αυτό το σήμα για τα βιολογικά προϊόντα, το ευρωπαϊκό σήμα. Άλλη μια ανησυχία μου είναι οι τροπολογίε που ψηφίστηκαν στην Επιτροπή ε, γεωργία που ζήτησαν να επανεισαχθούν οι προδιαγραφέ για την πώληση φρούτων και λαχανικών. Ε, όταν τόσα πολλά προϊόντα θέλουμε να μπορούν να απολούνται απευθεία στον καταναλωτή. Και αυτά απεσύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι. Υποστήριξα αυτή την κίνηση τότε. Α αφήσουμε την αγορά να θέσει τα πρότυπά τη και γι' αυτό θα ήθελα να παροτρύνω να υποστηρίξουν συνάδελφοι τη τροπολογική ομάδα μου και άλλων ομάδων που είναι σαφέστατε, είναι απλέ, να διαγραφούν αυτά τα στοιχεία από, την, από το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Ο κύριος Λορέντζο Φοντάνο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, επίτροποι κύριε Τσόλου. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μόλις ακούστηκαν και θα ευχαριστήσω και τον κύριο Σκοτά για το πολύ ευαίσθητο έργο που επετέλεσε όσον αφορά τη σχετική αυτή σημαντική έκθεση. Πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή που θα ψηφιστεί αύριο θέλουμε να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε τις, τα τυπικά προϊόντα κάθε περιοχής και χώρας Ευρωπαϊκής Ενώσεω και να τα αξιοποιήσουμε. Εγώ είμαι από την Ιταλία, μια χώρα που έχει 4.500 τέτοιου είδου προϊόντα και είναι ένας πλούτος της χώρας μας που δεν, θέλ, που θέλουμε να διαφυλάξουμε. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ο δρόμος για την αριστεία είναι ακόμα μακρύς, αλλά το μήνυμα που θα πρέπει να περάσει είναι ότι μόνο με την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων οι γεωργοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν με πολύ καλά και στην ε, παγκόσμια αγορά. Ε, λαμβάνοντα υπόψη και την κρίση, τη γενική κρίση που δυστυχώ ζούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παρά να υποστηρίξουμε την ποιότητα και την ανιχνευσιμότητα και τη διαφάνεια τη ενημέρωση όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα. Ε, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανεί τι είδου κατεργασία έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε καλλιέργεια και από πού προέρχεται το κάθε προϊόν. Και είναι και σωστό οι καταναλωτέ να γνωρίζουν αν τρώνε ένα μήλο που καλλιεργήθηκε παραδείγματο χάρη στη Βερόνα, στην περιοχή μου ή στην περιοχή του Βένετο και κατά τη διάρκεια αλυσίδα τη παραγωγική έχουν γίνει σεβαστέ οι επιταγέ τη κοινότητα, εάν τρώνε ένα μήλο που παράχθηκε στην Κίνα, παραδείγματο χάρη, που το μόνο που ξέρουμε είναι πω συχνά δεν έχουν τηρήσει εκεί και πόρα απέχουν από τι ε, πρακτικέ που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι γεωργοί. Ευχαριστώ. Σειρά τη κυρία Διάν Ντότ για 1,5 λεπτό. Uh, President... Πρόεδρε, Επίτροπε, σα ευχαριστώ που δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Οι καταναλωτές δικαίω ζητούν το φαΐ που αγοράζουν να είναι σύμφωνα με ψηλά ε, πρότυπα και ανοιχνεύσιμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να προωθηθούν αυτά τα πρότυπα και να γίνουν παντού αποδεκτά σε όλους τους ε, καταναλωτές προφανώς η πρόθεση και το marketing θα είναι εκείνη τα οποία θα βασιστεί η αποτυχία, επιτυχία του συστήματος και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουμε δράσεις κατά την απομιμήσεων ή των προϊόντων που δεν έχουν τις σωστές ετικέτες όπως πολλοί συνάδελφοι εδώ είμαστε κατά ενός ε, σήματος ευρωπαϊκού, ενός, ενός λόγου ευρωπαϊκού γιατί δεν θα έχει πολύ νόημα και δεν θα βοηθήσει πολύ τους κατανοτής. Ε, ονομασία προελεύσεως και γεωργικές ενδείξεις είναι πάρα πολύ γιατί προωθούν ε, την ε, τοπική παράδοση και προστατεύουν περιοχές που προωθούν την παραγωγή κάποιου συγκεκριμένου προϊόντα. Εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία είμαστε καθαρή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και γι' αυτό θέλω οποιοδήποτε σύστημα ακολουθεί να δημιουργεί ίσους όρους για όλους και ό,τι υιοθετηθεί δεν θα πρέπει να έχει αντίθετες επιπτώσεις σε χώρες όπως τη δικιά μου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι καλό να προωθήσουμε τα συστήματα εγγύησης των ποιότητων, της ποιότητας και της τοπικής πρόεδρευση. Ευχαριστώ, ρε Πρόεδρος. κυρία Κώστινγκερ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ε, θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την παραγωγή προϊόντων υψηλή ε, πρόεδρευση. Ένα συσχετισμό μεταξύ τη πρόεδρευση των προϊόντων και της ποιότητας του τροφίμου είναι απαραίτητη. Γι' αυτό υπάρχουν εδώ πολλές ευκαιρίες για τους παραγωγούς. Η ποιότητα σαν ε, παράγοντας κλειδί, έχει σε όλη την τροφιμική σημαντική ε, επίδραση. Ιδίως η παραγωγή προϊόν, τροφίμων υψηλής ποιότητας έχει παράδοση και είναι πολλές φορές η μόνη δυνατότητα ε, οικονομικές δραστηριότητες σε περιοχές ε, της Ευρώπης. Για να διατηρήσουμε την ποιότητα αυτή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ελέγχους και αντικειμενικά κριτήρια. Από την άλλη μεριά, οι οικονομικές σκέψεις ε, των ε, καταναλωτών παίζουν επίσης ένα ρόλο, γιατί η ποιότητα έχει τη τιμή της και οι παραγωγοί χρειάζονται ένα εισόδημα. Καμιά φορά ο, ο παίρνει το φθηνότερο, παρόλο που δεν είναι τόσο υψηλή ποιότητας. Αυτό που είναι σαφές ότι θα πρέπει να μπορεί ο καταναλωτή να επιλέξει βάσει σε, συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης χρειαζόμαστε γεωγραφικές ενδείξεις και ένδειξη προέλευσης. Χρειαζόμαστε μια προστιθε... προστατευόμενη σήμανση για τα προϊόντα αυτά από τις συγκεκριμένες περιφέρειες. Χρειαζόμαστε επίσης κάποια σήμανση για την οικολογική παραγωγή και για τα παραδοσιακά προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κύριος Δικάστρο. 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ξεκινά μια νέα φάση προβληματισμού στην Ευρώπη όσον αφορά την ποιότητα, που εννοείται όχι μόνο σαν στοιχείο που εγγυάται την ποιότητα στον καταναλωτή, αλλά ε, μπορούν να είναι, είναι ένα μοχλό που επιτρέπει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στου παραγωγού μα, όσο αυξάνεται και ο ανταγωνισμό στο παγκόσμιο σκηνή. Οι επιχειρήσει μα θα πρέπει να, να, να δουν να αναγνωρίζονται διακριτικά και ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων του, ε, αυτό που συνοδεύει δηλαδή την προσφορά του. Γι' αυτό, όπω αναφέρεται και στην έκθεση Σκοτά, τον οποίο ευχαριστώ τον κ. Σκοτά για την έκθεσή του, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προόδου για να εγγυηθούμε περισσότερε πληροφορίε που διατίθενται όσον αφορά την προέλευση, τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων παραγωγικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα είναι θεμελιώδε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να μπορεί να επιτρέπει στι οργανώσει που προστατεύουν και προωθούν τα ποιοτικά προϊόντα να μπορούν να προγραμματίζουν την παραγωγική προσφορά και να χρησιμοποιούν το δυναμικό παραγωγής και να προσαρμόζεται αυτό στις απαιτήσεις αγοράς βάσει ισοτήμων και μη διακριτικών ε, συνθήκων. Θέλουμε λοιπόν ε, ε, να καθαγιαστεί η ποιότητα μέσω αυτής της εκθέσεως σαν άξονας που προωθεί τη στρατηγική της Ευρώπης για τον τομέα τη ιερική παραγωγής και θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτάσεις τη Επιτροπής μας ούτω ώστε ένα από τα βασικά ισχυρά σημεία τη Ευρωπαϊκής Γεωργίας να μπορεί να μεταμορφωθεί σε πολύτιμο ανταγωνιστικό όφελος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντεκάστρο, ο κύριος Άγνιου έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, έχω συμφέρον ο ίδιος ως Γεωργός οι ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται και να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές. Είναι βασικό. Η κρίση έδειξε ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο πλήγει η βιομηχανία του. Απαγορεύσεις γίνονται αλλά για ορισμένε μόνο χώρες όχι για τη Ρουμανία, για την Βουλγαρία που έχουν ασυλία όσον αφορά τις αγωγές τους. Οι χώρες αυτές μπορούν να εξάγουν αυγά από όρνηθες σε κλοβούς με αποτέλεσμα άλλες χώρες να πλήττονται και ο ανταγωνισμός να γίνεται σε βάρος ε, ορισμένων μόνο χωρών από χώρες που μπορούν να πούν πολύ πιο φτηνά. Πρώτον λοιπόν αυτά τα ε, προϊόντα να λέμε ότι είναι εισαγόμενα και δεύτερον ε, καλύτερα αν μπορούν να απαγορευτούν άμεσα. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι ο καταναλωτής θα έχει την επιλογή. Ο κύριος Νταντάν τώρα. Για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, πιστεύω συμβολικό ότι είναι κύριε Επίτροπε που στην πρώτη σας παρέμβαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλήσατε ακριβώς για την πολιτική ποιότητας. Συμφωνούμε, νομίζω, στην προσέγγιση μα όσον αφορά τα προϊόντα ποιότητα. Αποτελούν μια ευκαιρία για τις πιο ευάλωτε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να βοηθήσουν τις περιοχές ε, αυτές, τον κόσμο που ζει εκεί, τους γεωργούς ιδιαίτερα. Όντω αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τον Ευρωπαίο καταναλωτή η ποιότητα, αλλά και προ τον καταναλωτή ολόκληρου του κόσμου το ζαμπόν από την Πάρμα, τα γαλλικά κρασιά, άλλα πρωτηριά της Ισπανίας είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η έκθεση που θα εγκρίνουμε αύριο δίχως άλλο προτείνει περισσότερη φιλοδοξία για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας που καθορίζονται ε, βάσει σημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περισσότερο ορατή, να φαίνεται και να φροντίσουμε να μην περάσει αυτό που θέλουν ε, οι μεγάλοι όμιλοι που θέλουν να εμποδίσουν τέτοια προϊόντα μικρής κλίμακας. Εγώ θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στην ε, ανάγκη που υπάρχει τη διαχείριση των προϊόντων να την έχουν οι που έχουν να κάνουν ε, με την προέλευση. Είναι πολύ βασικό για τα προϊόντα ποιότητας. Εξάλλου, η δικιά Επιτροπή υπερψήφισε περίπου ομόφωνα με τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θέλω να πω στους Βρετανούς για το άρθρο 19 που αφορά τα απορροκυπευτικά. Ναι συνάδελφοι, δεν θέλουμε να πάμε πίσω, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά ούτε και θέλουμε να δεχτούμε την πολιτική που προτείνουν αυτοί για τα απορροκυπευτικά που έχει σαν αποτέλεσμα διανομής να είναι η κύριοι του παιχνιδιού. Προσοχή λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν άλλο μέσο δρόμο. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να μας πείσετε για τον ενθουσιασμό σας υπέρ της ε, ποιότητας και γι' αυτό προτείνετε έμας ένα καλό κείμενο και γρήγορα. Έχουμε εμπιστοσύνη σε σας. Η κυρία Γκαρσία Πέρες τώρα. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων είναι βασικός παράγοντας στην διατροφική αλυσίδα και αποτελεί σημαντικό κρίκο επίσης υπέρ της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων γεωργών. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση Σκότα, όπου αναφέρονται και άλλα στοιχεία ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της στην ε, ανάπτυξη της ε, πολιτικής αυτής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δέσμευση από τους αγρότες μας για ποιότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό για τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωγραφική ένδειξη, οι αγορές, οι διμερείς συμφωνίες πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη τους. Η ολοκληρωμένη παραγωγή επίσης θα ευαισθητοποιήσει την παραγωγή ποιότητα σε όλες τις χώρες μέλη. Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανισορροπίες που υπάρχουν στην αλυσίδα εμπορίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προδιαγραφές εμπορίας ανατομέα και ενέχουμε κατευθυντήριε γραμμές από την Ευρώπη για καλή πρακτική όσον αφορά τα συστήματα που συνδέουν την ποιότητα των ε, γεωργικών προϊόντων και την αμοιβαία αναγνώρισή του. Θέλω έλεγχο των συστημάτων ιδιωτική πιστοποίηση που πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν απέτηση για να μπορέσουν να φτάσουν τα γεωργικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία Πέρες. Ο κύριος Σόν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Votre micro, ξεκινώ από την αρχή, λέει ο κύριος Σόινι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε περί τίνος πρόκειται αυτό που συζητούμε. Η οικογενειακή εκμετάλλευση είναι τοπικό τρόπο δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δημιουργεί τοπική ντόπια οικονομία. Είναι πολύ ανθρώπινη η οικογενειακή επιχείρηση όσον αφορά την προστασία των ζώων κλπ. Η ποιότητα των αγαθών είναι αυτό που δίνει στην ευρωπαϊκή οικονομία μια όθηση. Και η προέλευση του προϊόντος είναι πολύ σημαντική. Οι τοπικές ειδικότητες, οι τοπικές παραδόσεις είναι πολύτιμα πράγματα. Στη Φιλανδία, στη χώρα μου, έχουμε εξαιρετικό, εξαιρετικά προϊόντα έγια, κατσικίσιο, τυρί. Ε, είναι παραδοσιακά προϊόντα με μακρές ε, παραδόσεις και θα πρέπει να κατακτήσουν μερίδιο στην αγορά. Και τώρα με τον νέο επίτροπο θα πρέπει να μπορέσει ο κοινό επίτροπος να, ε, να φροντίσει να σκούνται αγροτικές δραστηριότητες παντού στην Ευρώπη. Να το θυμόμαστε. Αν το θυμόμαστε αυτό θα είναι έξοχο το μέλλον, διότι θα έχουμε καθαρά και πολύ ποιοτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά επόμενος ομιλητής, ο κ. Γιάρ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον εισήγητη για την τόσο καλή του έκθεση. Πραγματικά είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία τα εργατικά προϊόντα υψηλής ποιότητας για να μπορούν να επικρατήσουν στον διεθνή αγορά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αγροτικά αυτά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη σήμερα τηρούν υψηλά ποιοτικά πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θεωρούνται διεθνώ υψηλά αυτό δεν το ξέρουν όλοι ακόμα και αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ποιοτική της πολιτική και την πολιτική της ενημέρωσης γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο που το οι παραγωγείς να κινηθούν ακόμα περισσότερο στον τομέα της τροφιμικής ασφάλειας και της ποιότητας των εργατικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι κανένας θα πρέπει να τρώει τα αγροτικά προϊόντα αυτά χωρίς πρόβλημα. Μια σήμαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια υποχρεωτική περιφερειακή γεωγραφική ανάπτυξη, ε, συγγνώμη, δεν αποκλείονται το ένα από το άλλο. Από την άλλη μεριά όταν πρόκειται για το μέγεθος των ε, ε, συσκευασιών και τη μορφή των προϊόντων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ορίζει πόσο μεγάλη μια, μια πίτσα ή ε, πόσο στραβή είναι μια μπανάνα. Αυτό που προέχει είναι η ποιότητα. Γιατί αν θέλει κανένας ένα βιομηχανικό προϊόν μπορεί να, επιμείνει να είναι ε, πάντα του ιδίου βάρους του ίδιου μορφής. Γι' αυτό εμείς ε, όμως βασιζόμαστε στην ε, ποιότητα και όχι στην, στο ενιαίο της συσκευασία. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και βασιζόμαστε στην, ε, στο Κοινοβούλιο και στον Επίτροπο κ. Η κυρία ε, Νταντσίλα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την προσέγγιση του, του τόσο σημαντικού αυτού θέματο τη ποιότητα των ιδιωτικών προϊόντων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας απασχολεί ιδίω η υγεία, η ασφάλεια και η τροφιμική αξία των προϊόντων. Οι καταναλωτέ επίση είναι όσο πάει και πιο προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο ε, η Γεωργία συμβάλλει στην ποικιλομορφία, στην ε, σταθερότητα των, ε, του κλίματος και ούτω καθεξής. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ ενδιαφέρονται κυρίως για την ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλεονέκτημα με την ποιότητα που οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε όλη την τροφιμική αλυσίδα στην οποία συμβάλλουν και οι παραγωγοί και οι καταναλωτέ. Υπάρχουν όμως ορισμένες πτυχές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα. Θα πρέπει η Ένωση να προωθεί τα ποιοτικά προϊόντα και να τα προστατεύει και διεθνώς. Και στο ίδιο σκεπτικό πιστεύω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε πιο αυστηρούς ελέγχους για τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Γιατί αυτό θα επιτρέψει έτσι ίσες ευκαιρίες για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Ε, Ευχαριστώ, κύριο Ντανέλη, σε ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα για τον καταναλωτή μέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας για τον παραγωγό και μέσω ενίσχυσης της περιοχής παραγωγής τους. Γι' αυτό και επιδιώκεται η κατοχύρωσή της, μεταξύ άλλων και με τη σήμανση. Σήμερα όμως η κοινοτική νομοθεσία περιορίζει την υποχρεωτική σήμανση του τόπου παραγωγής μόνο σε ορισμένα προϊόντα εξασφαλίζοντας τους ειδική μεταχείριση αφήνοντας έξω γεωργικά προϊόντα μεγάλης διατροφικής αξίας και προτεραιότητας για τον καταναλωτή. καλούμε λοιπόν το κοινοβούλιο να υιοθετήσει πιο συνεπή και λογική στάση υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων του καταναλωτή προκρίνοντας την υποχρεωτική σήμανση του τόπου παραγωγής για όλα τα γεωργικά προϊόντα συμπεριλαμβάνοντας και τα μεταποιημένα προϊόντα με ένα μόνο συστατικό όπως παραδείγματος χάρη είναι το γάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Όποιον πάρει το μάτι της πρόεδρο. Κύριος Νικουλέσκου. Πρώτα, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι πολιτικές στο θέμα ποιότητας αγροτικών προϊόντων είναι μία λύση για πολλές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει όντως να τονίζουμε την ποιότητα και όχι την ποσότητα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μακροπρόθεσμα κέρδα. Χρειάζεται λοιπόν συνεκτική πολιτική σε αυτό το τομέα, κάτι που προσφέρει στους Ευρωπαίους γεωργούς να είναι ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές. Η έκθεση Σκότα είναι πολύ καλή και οι προθέσεις του Επιτρόπου είναι επίσης καλές ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, για την ποιότητα. Χρειαζόμαστε όμως και κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική για το μέλλον που να χρηματοδοτείται επαρκώς με προϊόντα ποιότητας και με μεγαλύτερο προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Χρειαζόμαστε τα μέσα, τα εργαλεία που πρέπει να έχουμε για να ενισχύσουμε την ποιότητα αλλά και να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στι ανατολικέ και δυτικέ χώρε. Η κυρία Μέμερτς τώρα. Ένα λεπτό. στη συζήτηση για την ποιότητα και την υπολογιστική σήμαση των ε, γεωργικών προϊόντων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιτικέ ε, αποφάσει θα πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμε. Στι τροπολογίε 4 και 5 δεν βλέπω να είναι πρακτικά εφαρμόσιμε και αυτό θα σα απορρίψω. Η σήμαση ποιότητας ε, είναι θετική εάν είναι εθελοντική. Γιατί αυτό δεν είναι δυνατό του προβού να είναι επιτυχή στι αγορέ. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένα ε, θελοντικά ε, σήματα επιβάλλονται και θεωρούνται σήματα ποιότητας πράγμα που περιορίζει την δυνατότητα επιλογής ε, των παραγωγών. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό της, γεωγραφική της γεωγραφικής προέλευσης παραδείγματος χάρη του γάλακτος. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, η καλή θέληση να μην οδηγήσει σε τεράστια γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Pardonnez-moi d'avoir votre nom. <laughs> E, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο νέα της εκθέσεως. Εκεί τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί κάποια συμφωνία όσον αφορά τη, τις συνθήκες πωλήσεως που να ισχύουν για όλα τα προϊόντα και να υπάρχουν και να πληρούνται οι προδιαγραφές για την προστασία των ζώων κλπ. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι πρέπει να εφαρμόζονται ίδιες προδιαγραφές στα δικά μας προϊόντα και στα προϊόντα των άλλων. Δυστυχώς η φωνή μας δεν έχει εισακουστεί. Αποτέλεσμα αυτού, οι γεωργοί μας και οι μεταποιητές μας να έχουν μεγαλύτερο κόστος. Και είναι αθέμητος έτσι ανταγωνισμός. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και εκτιμώ λοιπόν αυτά που τονίζονται σχετικά με το θέμα στην έκθεση. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. Η έλεγχη των ε, τροφίμων είναι ουτοπία και οι επιπτώσεις επίσης. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα όταν υπάρχει μήνες κίνδυνος ασθένειας θα μπορούσαν οι υπηρεσίε να προειδοποιήσουν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να το κάνουν και αυτό οδηγεί σε όλε τι κρίσεις που γνωρίζουμε. Πολλέ φορές οι ελεγκτές των τροφίμων έχουν πρόβλημα με την ελληματική σήμανση και το ίδιο ισχύει για τους καταναλωτές. Λέει α πούμε ε, παραγωγός ενώ έχει παραχθεί στην ε, ε, βιομηχανία ή λέει ότι προέρχεται από την Αυστρία ενώ τα, οι πρώτες ύλε έχουν προέρχεται από όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να πούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε έτσι όταν έχουμε τόσους που δεν ακολουθούν την σωστή άγουσα. Και αν μόνο οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν τις διαδικασίε αυτές και όχι οι μεγάλες, τότε είναι το πρόβλημα τεράστιο. Ευχαριστώ κύριε Στόρπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε σήμερα ότι αυτά τα προϊόντα που έχουν την ονομασία προέλευσης είναι στο επίκεντρο. έχετε δίκιο και αυτό ισχύει για προϊόντα που παράγονται κάτω από δύσκολε προποθέσει, παραδείγματο χάρη σε ορεινέ περιοχές και γι' αυτό χρειάζονται μεγαλύτερα περιθώρια ε, κέρδου. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα η παραγωγή να οργανώνονται σε επιτροπές προστασίας. Αυτό δεν είναι αντίθετο με τον ανταγωνισμό και αν είναι αντίθετο είναι πολύ μικρότερο το πρόβλημα από ότι με τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. Δεν θέλω να πω δύο λόγια όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητα. Δεν γνωρίζω τι συζητήσει στον τύπο ξέρω ποιες είναι οι συζητήσεις για τα ίσια ή τα στραβά αγκούρια. Όμως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί είναι στοιχεία που επίσης χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Φερέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, οι μηχανισμοί πιστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν ε, στην αναβάθμιση της δουλειάς ε, των ε, εργαζομένων, των γεωργών, να αυξηθεί ο μισθός τους, για παράδειγμα, τα εισοδήματά τους. Από την άλλη μεριά, οι διαδικασίες πιστοποίησης καθυστερούν, είναι περίπλοκες και πλήττουν άμεσα τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το κόστος παραγωγής και μια κατανομή της αλυσίδας πλήττει ακόμα περισσότερο τον παραγωγό. Αν υπάρχουν περισσότεροι ενδιάμεσοι που πρέπει και αυτοί να κερδίσουν κάτι, οι παραγωγοί παίρνουν ακόμα λιγότερα. Και η ασφάλεια των καταναλωτών περνάει από μια πιστοποίηση από δημόσιες αρχές και όχι από τον παραγωγό ώστε να του κοστίζει ακόμα περισσότερο η παραγωγή του. Χρειάζεται επίσης μια μεταρρύθμιση σε βάθος της κοινή γεωργικής πολιτικής και να υπάρχει δικαίωμα κυριαρχίας στην παραγωγή τροφίμων. Δυστυχώς η απορρίθμιση σε διεθνέ επίπεδο έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους παραγωγούς, όπως επίσης και οι συνθήκες στην αγορά, κλπ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν αξία στην παγκόσμια αγορά λόγω της ποιότητάς τους. Συζητάμε τις μελλοντικές προοπτικές των, της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες, διότι πλεονεκτούμε εκεί σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι κάτι σημαντικό και για την τοπική κοινωνική ζωή. Θα πρέπει η ποιότητα να υποστηριχθεί και να υπάρχει και στην ετικετοθεσία μεγαλύτερη σαφήνεια για να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει. Και έτσι θα προστατεύουμε την ποιοτική παραγωγή ε, γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει να φαίνονται και ποια προϊόντα περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και γενετικά τροποποιημένες ε, πατάτες, παραδείγματος χάρη, κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για να μην απειλείται η υγεία μας αν λείπουν τέτοιοι σαφείς κανόνες όσον αφορά αυτά τα προϊόντα. Επόμενος, ο μιλητής, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, χάρη στην κοινή αγροτική πολιτική έχουμε ποιοτικά προϊόντα στην Ευρώπη, προϊόντα υψηλής ποιότητας και χρειάζεται η σωστή ποιότητα και η σωστή παροχή αυτών των προϊόντων που εξασφαλίζει την επιστημιστική ασφάλεια οι πληροφορίες για την ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει ε, να φτάνουν στον καταναλωτή. Και τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά, στην Ευρώπη, θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Όλα λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία. Διότι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά καθορίζουν την ποιότητα και η περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλη των πρώτων υλών και το, ο τόπος μεταπή πρέπει να αναφέρεται για να ξέρει ο καταναλωτής ακριβώς τι αγοράζει και τι πράγμα πληρώνει. Ε, αυτό θα είναι κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Εν συγκρίση με τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν θα πληρούν τα ίδια κριτήρια. Η επιτυχή έκθεση του κ. Σκοτά είναι πραγματικά προ όφελο τη προστασία του καταναλωτή. Γιατί πρέπει τα ε, γεωργικά προϊόντα να είναι υψηλής ποιότητα και να μην απειλούν την υγεία των καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι καλό να βελτιώσουμε την ε, σήμαση ονομασία προέλευσης των αγροτικό προϊόντο. Για κάθε αγροτικό προϊόντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει η ονόμαση προέλευση. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει ε, απάτη. Παραδείγματο χάρη έρχονται κάποια ζώα από άλλες χώρες ε, στην ε, Αυστρία και χρησιμοποιούνται μετά για αυστριακά προϊόντα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Θα πρέπει η τοπική παραγωγή να ενισχύονται προς όφελο των ε, παραγωγών και των γεωργών. Ευχαριστώ. Ο τελευταίο ομιλής είναι η κυρία Ντετέλτσεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρω τον συνάδελφο Σκοτά για την έκθεσή του, η οποία αναφέρει σαφώς τη βούληση που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις τις σχετικές με την κοινή αγροτική πολιτική. Υποστηρίζω ένθερμα το θέμα της ευρωπαϊκής ετικέτας, του ευρωπαϊκού σήματος, που θα δείχνει ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί στην Ευρώπη. Όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης, να είναι υποχρεωτική αν το κάνουμε αυτό, προστατεύουμε την παραγωγή διαφόρων περιοχών και παρέχουμε τα αναγκαία χέγγια στον καταναλωτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το μέσο που προστατεύει τα παραδοσιακά προϊόντα. Δεν είναι κακό να ξέρει κανείς ότι η φέτα είναι παραγωγή της ε, Ελλάδας και ένα άλλο τυρί ε, παράγεται στη Βουλγαρία. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων και έτσι την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ, λίγο. Πρόεδρο. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε, μετά από αυτές τις πολλές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα όλες τις ε, ερωτήσεις και τα σχόλια. Δεν θα απαντήσω ε, στο καθένα χωριστά, αλλά θα απαντήσω συγκεντρωμένα στις σα για τη συγχώνευση των διάφορων συστημάτων γεωγραφική ένδειξη. Καταλαβαίνω τι ανησυχίε ορισμένων ευρωβουλευτών. Σα ε, διαβεβαιώ όμω ότι στόχο μου δεν είναι να καταστρέψω κάτι που λειτουργεί καλά. Που δεν θέλω να καταστρέψω κάτι το οποίο αρέσει στους καταναλωτές. Θέλω όμως να υπάρχει περισσότερη συνοχή στο σύστημα προστασίας της ποιότητας Ιδιαίτερα μάλιστα που προσπαθούμε στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων να αναγνωριστεί αυτό το σύστημα. Άρα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να μπορούν οι εταίροι μας να το κατανοήσουν. Δεν σκοπεύω λοιπόν έτσι για την... Ε, να συγχωνεύσω για να συγχωνεύσω χωρί λόγο. Όχι. Δεν θέλω να πειράξω πράγματα τα οποία γνωρίζει καλά ο καταναλωτή και τα θέλει και τον εξυπηρετούν. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητα. Και εδώ πρέπει να το συζητήσουμε, να δούμε τι στόχους θέλουμε να πετύχουμε από ένα τέτοιο λογότυπο. Γιατί αν πρόκειται μόνο για να φαίνεται ότι τηρούνται οι βασικές αρχές που όλοι οι Ευρωπαίοι γεωργοί τηρούν και ότι τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν τις ίδιες αυτές προδιαγραφές γιατί προσοχή όλα τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα πρέπει να τηρούν ε, τους, ε, τις ελάχιστες προδιαγραφές ε, υγειονομική προστασίας. Ποιο είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσουμε τα δικά μας προϊόντα από τα άλλα. Χρειάζεται ένα λογότυπο Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να μιλάμε για τον τόπο παραγωγής, προέλευσης. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο καλύτερος μηχανισμός. Το σκεφτόμαστε. Για τι γεωγραφικέ ενδείξει, τώρα σε διεθνέ επίπεδο. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι κάτι που θέλω να φροντίσω, γιατί θέλω να αναγνωρίσουν το σύστημα οι εταίροι μας διεθνώς και το προσπαθούμε αυτό στα πλαίσια του ΠΟΕ, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε και κάθε φορά που έχουμε τη δυνατότητα και διμερώς σε διμερείς συμφωνίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και επιπλέον κατά τη διάρκεια της θητείας μου θέλω να ενισχύσω την πολιτική επικοινωνίας και ε, πρόθεσης του Ευρωπαϊκού Σήματος ποιότητας. Γιατί η ποιότητα αποτελεί ένα ατού για μας στη διεθνή σκηνή. Όσον αφορά τώρα τις ορεινές ε, περιοχές, ε, προέλευση δηλαδή ορεινή, νησιώτικη κλπ. Και εδώ πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φορτώνουμε με παραπάνω δουλειά τους παραγωγούς. Να είναι ίσως εθελοντική βάση. Όσον αφορά τώρα τις διαπαγγελματικές οργανώσεις και το ρόλο τους στην διαχείριση των γεωγραφικών ε, ενδείξεων, έχουμε προβλέψει όσον αφορά το γάλα, ιδιαίτερα γιατί εκεί επικεντρώνεται το θέμα, προβλέψαμε μελέτη για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του τέλους των ποσοστώσεων στη λειτουργία του συστήματος αυτού προστασίας ποιότητας. Ελπίζω βάσει της μελέτης αυτής να καταλήξουμε και σε συμπεράσματα για τα μέτρα που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο συγκητής τώρα έχει το λόγο, ο κύριος Σκοτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Τσόλος. Εγώ θα μιλήσω για τη γη. Πολύ σύντομα, στη γη παράγουμε τα προϊόντα μας. Ε, αυτή πρέπει να συντηρήσουμε για το μέλλον και για τους άλλους που θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν. Από μια απλή σκέψη τέτοια λοιπόν θα πέναγα στον παραγωγό, εκείνο που επεξεργάζεται τη γη, χρησιμοποιεί τη γη και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με εκείνο που μετά θα χρησιμοποιήσει το προϊόν, το εμπορικό προϊόν που θα βρει στην υπεραγορά, στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αγοράσει. Είναι σωστό να σεβαστούμε πάνω απ' όλα τη γη που παράγει το προϊόν τον ενδεχόμενο μεταπητή, αλλά πάνω απ' όλα τον καταναλωτή. Και για τον καταναλωτή, εγώ θα έκανα μια πρόταση. Δεν ξέρω αν θέλει να τη δεχτεί κάποιο, γιατί δεν ζητάμε από τον καταναλωτή τι θέλει να ξέρει. Και έτσι θα ξέρουμε ποια θα πρέπει να είναι η ετικέτα που θα μπορεί να διαβάσει, να καταλάβει ο καταναλωτή απλουστεύοντά την ενδεχομένω σε συγκρίση με τι πολύ περίπλοκες ετικέτε που έχουμε σήμερα. Γιατί να μην ξέρει ο καταναλωτή ότι μπορεί να αγοράσει ένα λίτρο ευρωπαϊκού γάλακτος ή κάποιο, ένα λίτρο γάλακτος που έρχεται από τη Βραζιλία. Αυτός μπορεί να κρίνει το βραζιλιάνικο γάλα είναι καλύτερο από αυτό της ευρωπαϊκής κοινότητας. Όμως ελπίζω αυτή η έκθεση να είναι χρήσιμη ούτω ώστε και ο Τσόλος να μας δώσει αργότερα κάποιες λεπτομέρειες για να αναπτυχθεί αυτή η αλυσίδα που είπα, γη, παραγωγό, ενδεχόμενο μεταπητή και καταναλωτή. Ασφάλεια στην αλυσίδα και μέσα στην ασφάλεια και ποιότητα που την ανέφεραν όλοι και όλοι είμαστε υπέρ της αυξήσεως της ποιότητας του προϊόντος μας για ε, να μπορούμε να τρώμε καλά και να τρώμε υγιεινά για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ποιότητα και το προϊόντος αλλά της παρέμβασής σας. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο. Πάμε στην επόμενη συζήτηση. Τη δήλωση της Επιτροπής